την Ισιαρή ότι έχουμε λάβει κατάλογο για ε, ονόματα που θα συμμετέχουν στις επιτροπές και διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις ε, θα επικυρωθούν αυτές οι